ως ένα από τα αρχαιότερα μέλη αυτού του Κοινοβουλίου και θέλω να σας πω ότι αν φύγετε ε, θα μου λείψετε. Αλλά θέλω να υπογραμμίσω το αν, αν, το υπογραμμίζω αυτό το αν φύγετε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Η κυρία Σκοτ Κέιτο, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το Σαββατοκύριακο η Πρωθυπουργό ε, προσπάθησε να βρει κάποια λύση για το deal. Θέλησε να διαπραγματευτεί με όλους εκείνους οι οποίοι είναι όμως η μειονότητα της μειονότητας στο κόμμα της. Και μπορούμε να φανταστούμε τι τους είπε. Ότι αυτή η διαδήλωση στο Λονδίνο ε, και οι υπογραφές για το άρθρο 50 αυτά καταδεικνύουν ότι η χώρα είναι ε, κατά του Brexit. Ψηφίστε λοιπόν τώρα, αλλιώς θα χαθεί το Brexit. Ίσως να γίνουν πολλοί θέλουν και άλλες εκλογές. Αυτό όμως είναι τρόμος για τους τόρεις, γιατί αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εκφράσουν την άποψή τους και να δείξουν ότι είναι κατά του Brexit. Οι συντηρητικοί φοβούνται τη βούληση του λαού, αλλά εμείς δεν θα σιωπήσουμε. Στη χώρα μας αυξάνεται όλο και περισσότερο η αντίσταση κατά της, του Brexit. Ε, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι στην Ήπειρό μας ε, υπάρχει φιλοευρωπαϊσμός και ότι οι πολίτες, αν κληθούν θα ψηφίσουν υπέρ του να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,5 λεπτό η κυρία Άντερσον και αν αυτή είναι η τελευταία σου θα σας δώσω και άλλα 30 δευτερόλεπτα. Πριν από το δημοψήφισμα μας ε, είχαν πει ότι το Brexit θα επιφέρει τεράστια ζημιά στην Ιρλανδία. Και πράγματι αυτό ήταν σωστό. Εμείς κάναμε εκστρατεία έτσι ώστε ο Βοράς να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ε, ξέρουμε ποιες είναι οι ζημιές του Brexit, ε, τι θα επιφέρει στη δική μας, στο δικό μας το νησί. Και είχαμε δίκιο και το πιο σημαντικό, η πλειοψηφία των πολιτών στην Βόρεια Ιρλανδία συμφώνησαν με μας. Όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μας προειδοποίησαν ε, όλους ε, σχετικά με την τακτική των Βρετανών και θέλω να σας πω ότι ε, θα σας αφήσω να κρίνετε μόνοι σας το πόσο δίκιο είχαμε. Η άγνοιά τους και η έπαρση τους που στηρίχθηκε και από το κόμμα DUP μας έφερε στην Άβυσσο, στο χείλος της Αβύσσου και εκεί βρισκόμαστε ακριβώς τώρα. Το Brexit περιγράφεται ως ε, μια σειρά από αναπάντητα ερωτηματικά. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα το οποίο υπερισχύει και το οποίο κατ' ουσίαν ε, συνεπάγεται και μια πολύ απλή απάντηση για την Ιρλανδία και ίσως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να βρούμε από αυτό το απόλυτο χάος. Η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ε, που στηρίζεται από πάρα πολλούς παρευρισκόμενους είναι εκείνη που περιλαμβάνει τη λύση. Κύριε Τούσκ, σας καλώ να βασιστείτε στην δήλωση του Συμβουλίου της, ε, του Απριλίου του 2017, να συνεχίσετε τις απαραίτητες συζητήσεις και να απαντήσετε στα μεγάλα ερωτήματα, να αποδραματικοποιήσετε το θέμα, γιατί εάν απομακρύνουμε τα σύνορα θα απομακρύνουμε το πρόβλημα να υπάρχει πρόγραμμα για την ενότητα της Ιρλανδίας με βάση τη συνένεση. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Κύριος Πάξας ε, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι όλο και περισσότερο απομακρυνόμαστε από το πνεύμα της Ένωσης των Εθνών. Και τασόμαστε όλο και περισσότερο υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Αυτή είναι η νέα ιδεολογία και όλο το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό κατεστημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί παρά να ενδώσει σε αυτή την ιδεολογία. Τη πρόσπιση δηλαδή πάση θυσία των συμφερόντων των επιχειρήσεων και κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων ει βάρο των συνόρων των εθνών. Αυτή η παγκοσμιοποίηση έχει αρνητική επίπτωση και στο περιβάλλον και επίση ε, φτωχοποιεί τα έθνη και πλήττει το κράτος δικαίου. Οι πολίτες δεν νιώθουν πια να είναι σαν στο σπίτι τους, στην πατρίδα του. Ε, αλλά τα κράτη ιδιωτικοποιούνται από τις πολιτικές ελίτ, περιθωριοποιώντας τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίων απειλούνται από τη φτώχεια. Εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλώνουν σε οικογένειες που ζουν στο κατόφλι της φτώχειας. Θα πρέπει να αντισταθούμε σε μια τέτοια πολιτική και θα πρέπει να είμαστε κατά της παγκοσμιοποίησης και μάλιστα γρήγορα. Ο κύριος Μπέ για ένα λεπτό. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ορθώ στηλίτευσε σε συνέντευξη τύπου την αφέλεια των Ευρωπαίων στα εμπορικά θέματα. Αυτή τη στιγμή η αδιάβια του όμω δεν τον εμπόδισε να βάλει την υπογραφή του στα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ το κείμενο αυτό ήταν πολύ αντιφατικό. Αναφερόταν μάλιστα το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει τα συμφέροντά τη απέναντι σε αθέμητε πρακτικέ των τρίτων χωρών. Επίση, ε, ε, καλεί για πλήρη χρήση των εργαλείων τη ε, εμπορική άμυνα. Θαυμάσια. Το ίδιο όμω έγγραφο ρητά παροτρύνει να συναυθούν νέε εμπορικέ συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών και επίση επιβεβαιώνει την προσήλωσή του σε ένα ανοιχτό εμπορικό σύστημα και αντιστέκεται σε οποιαδήποτε μορφή προστατευτισμού, ε, λένε οι Ευρωπαίοι. Κάτι που ε, προκαλεί το γέλο στους Αμερικανούς και Κινέζους που σοριδών αγοράζουν τι επιχειρήσεις μας. Θα πρέπει λοιπόν να, σταθεί, να τεθεί ένα τέρμα ε, σε, αυτά, σε αυτές τις ψευδεστήσεις. Έχουμε κολλήσει στο παλιό δόγμα των ελεύθερων συναλλαγών, αλλά δεν είμαστε ένα προστατευμένος χώρος. Είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα που δεν έχουν κανένα κόμπλεξ, να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους και να προσπίσουν τις οικονομίες τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, για ένα λεπτό, κύριο Χούκεμ. Ε, νομίζω ε, ότι πολλές συγκρίσεις ε, ε, με την ιστορία μπορούν να γίνουν, δυσμενείς πάντοτε για την Πρωθυπουργό Μέη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς προσπαθεί να παρακάμψει τη βούληση των λαών. Ο λαός της Ευρώπης ε, αντιλαμβάνετε τις ανησυχίες. Αν ε, έχετε την αυταρέσκεια να πιστεύετε ότι μόνο για ψήφο διαμαρτυρίας ε, δέχτηκαν να αποχωρήσουν και ψήφισαν να αποχωρήσουν οι Βρετανοί, κάνετε λάθος. Ε, βλέπουν να ανοίγεται μπροστά τους μια νέα πολιτική. Το κοινοβούλιο αυτό ε, φοβάται την επέλαση του ευρωσκεπτικισμού. Ε, ε, όλα αυτά θα καταρριφθούν. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σταθώ στο θέμα του Brexit, αναλύθηκε εκτενώς. Ε, το Brexit ε, μας κρατάει σε ομοιρία, μας εμποδίζει να ατενίσουμε το μέλλον μας. Θα πρέπει να δούμε την ε, πολιτική αυτή κρίση ως πολιτική κρίση του Ηνωμένου Βασιλείου και οι επιχειρήσεις μας και οι πολίτες μας έχουν κουραστεί επιτέλους από αυτή την κολυσίεργεια. Θα πρέπει να ληφθεί επιτέλους μια απόφαση. Ξέρω ότι το Συμβούλιο ασχολήθηκε με την ε, ανάπτυξη και με το βιομηχανικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στη τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να καλύψουμε το χαμένο έδαφος στα θέματα του ψηφιακού κόσμου για να διαφυλάξουμε την θέση των Ευρωπαίων στην αμελλοντική οικονομία γιατί η Κίνα έχει λάβει πολύ σημαντική θέση και είναι επιτακτική ανάγκη της Ένωσης να υψώσει το παράδειγμα το παράστημά της. Χαίρομαι που η Γαλλία παίζει σημαντικό ρόλο, είναι κινητήριος μοχλός στα θέματα αυτά και υιοθετήσαμε ένα πιο ε, κατηγορηματικό τόνο. Ακόμη όμως υπάρχουν διχασμοί στο Συμβουλίο. Άκουσα ότι ο πρόεδρος Γιουνκέρ μας είπε ότι δεν θα πρέπει να είμαστε ανοιχτό ξαφαραγό αμπέλι, αλλά ανοιχτοί στο εμπόριο. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποβάλει φιλόδοξε προτάσει για το 2050. Βρισκόμαστε σε ολισθηρό έδαφος και φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη κοφεύουν σε αυτή την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν δράσεις. Πότε επιτέλου θα ξυπνήσουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροντρίγκε, για δύο λεπτά. Αγαπητή Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ερηνό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν τις ευρωεκλογέ. Και φυσικά περιμένουμε πολλά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πριν από 20 χρόνια καταφέραμε να προσδιορίσουμε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο για να δούμε την Ευρώπη στην παγκοσμιοποίηση ήταν το πρόγραμμα της Λισαβόνας και ακολούθησε η συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι και η ώρα να χαράξουμε ένα νέο μεγάλο επίβολο σχέδιο για την Ευρώπη και τον κόσμο, γιατί ο κόσμος μεταβάλλεται ραγδαίως. Η Κίνα σίγουρα είναι πολύ σημαντικό εταίρο και είναι σημαντικό να πούμε αυτά που είπαμε, ότι θέλουμε στρατηγική εταιρική σχέση με την Κίνα, αλλά αμφίδρομη, με σεβασμό και των δικών μας αξιών. Επίσης γνωρίζουμε ότι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και η προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα στο επόμενο πρόγραμμα εργασιών μας. Πολλό δε μάλλον όταν μιλούμε για την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Γνωρίζουμε ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να τη την ψηφιακή επανάσταση, να προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο διαχείρισης της ψηφιακής επανάστασης. Και αυτό θα πρέπει να πούμε στους Κινέζους εταίρους μας στην επερχόμενη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνα. Κίνας. Ευρωπαϊκός τρόπος ψηφιακής επανάστασης σημαίνει προστασία της ιδιωτικότητας, προστασία της ασφάλειας και προστασία της ελευθερίας. Επίσης σημαίνει χρησιμοποίηση των ψηφιακών εργαλείων όχι για να υπονομεύσουμε, αλλά για να εμπλουτίσουμε τη δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή επανάσταση θα πρέπει να βρεθεί στην καρδιά της πρόθεσης νέων αγαθών και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις ε, ανθρώπινες ανάγκες, στις ανάγκες των πολιτών. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για να έχουμε πιο σύγχρονα σύστημα, συστήματα πολιτικής προστασίας και να προστατεύσουμε τους πολίτες στη διάρκεια αυτής της ρηξικέλευτης επανάστασης. Ε, και πιστεύω ότι για τους Ευρωπαίους η γνώση, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, ε, αυτά είναι τα βασικά μας ατού. Και θα πρέπει αυτά να εμπνεύσουν και το είδος της τεχνητής νοημοσύνης που θέλουμε να αναπτύξουμε. Να, να δημιουργήσουμε λοιπόν, να εφεύρουμε τη νέα, τη νέα όψη του μέλλοντος. Γιατί υπάρχει πολύ φως μετά από αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι του Brexit, το σκοτεινό. Κύριε Μπιτσότο η Ευρώπη των μεταναστών και τις φορολογίες, η Ευρώπη του Γιούνκερ, της Μέρκελ και του Μακρόν. Αυτό είναι το τέρμα. Ε, οι Ιταλοί ε, στις 26 ε, Μαΐου θα στείλουν εσά στο σπίτι σας κύριε Γιούνκερ και τον Επίτροπο Φαστάγκερ που έκαναν ζημιά στους Ιταλούς. Εμείς με τον κύριο Σαλβίνη είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε από την κορυφή την Ευρώπη που είναι δούλη των τραπεζών. Εμείς θέλουμε να συστήσουμε μια νέα Ευρώπη. Μια Ευρώπη διαφορετική. Μια Ευρώπη που υπερασπίζεται τα σύνορα, που θα αναχαιτίζει την παράνομη μετανάστευση, που θα προστατεύει τους εργαζόμενους μας. Ε, κύριε Γιούγκερ και αγαπητοί γραφειοκράτες, όλα αυτά τα χρόνια προκαλέσατε καταστροφές, ταπεινώσατε τον Ιταλικό λαό, αλλά και άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Οι Ιταλοί με μεγάλη περηφάνεια, επιτέλους μετά από λίγες εβδομάδες θα σας στείλουν στο σπίτι σας. Εμείς από τη Λέγκα, από το κόμμα αυτό, ε, θα είμαστε το πρώτο κόμμα στην Ευρώπη, γιατί η δική μας η ψήφος, η ψήφος των πολιτών μας, θα είναι μια πραγματική ψήφος της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο κύριος Ουγιασδόφσκι για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τη συζήτηση για τον Brexit. Γιατί είναι συγκινησιακά φορτισμένη και χρησιμοποιείται μερικές φορές για εσωτερικούς ε, πολιτικούς λόγους. Και μάλιστα ο κύριος Φαράζ επέκρινε τη συνθήκη των Βερσαλιών ως ε, ταπεινωτική για τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό είναι πραγματικά ανοησία. Επανέρχομαι στο πρόγραμμα εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εκτιμώ ιδιαιτέρως ε, τα γεωπολιτικά συμπεράσματα και κυρίως ε, η διατήρηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και αν μιλούμε για την ουσιαστική αλληλεγγύη, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης. Η ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης είναι ασφάλεια ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τα οικονομικά θέματα και τα οικονομικά συμπεράσματα ή το θέμα της ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Το έγγραφο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου αναφέρει ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία ενιαίας αγοράς και στην άρση των εμποδίων που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των, της επιχειρηματικότητας. Βέβαια, μερικές φορές ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορθώνουμε εμπόρια ε, στην οικονομία και τέτοιο χαρακτήρα δημιουργία οικονομικών εμποδίων έχουν κάποιε ψηφοφορίες που θα κάνουμε για τις μεταφορές. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη λοιπόν ότι ε, δεν θα πρέπει να δημιουργούμε φραγμούς στην ε, οικονομική ελευθερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριο Γκονσάλε Πόν. Η συνάδελφος Εστέρ Ντελάνκε μα είπε πολύ σωστά ότι το Brexit συζητούμε, αλλά όλες οι βουλευτικές έδρε από τους του Brexit είναι κενές έρχονται απλώ για να εισπράξουν ε, την αμοιβή του όχι για να εργαστούν οι ευρωβουλευτέ που εκπροσωπούν ε, την τάση αυτή του Brexit. Ενώ εκατομμύρια φορολογούμενοι πληρώνουν του μισθού του. Θα πρέπει επίση ε, να αποφασίσουν μια για πάντα, μέσα ή έξω. Τρίτη λύση δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει δυνατότητα να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο και αν δεν σκέφτονται κάτι τέτοιο στο μέλλον, τότε δεν θα πρέπει να ξαναγίνουν ευρωεκλογέ. Αν είναι μόνο για να συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει, εδώ δεν είχαμε ε, βουλευτές από τον Καναδά όταν συζητήσαμε τη συμφωνία με τον Καναδά, ούτε ε, βουλευτές από την Ιαπωνία όταν συζητήσαμε την εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία. Γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε Βρετανούς ε, βουλευτές για να συζητήσουμε εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως δεν έχουμε Ισπανούς, Γάλλους βουλευτές στην Βουλή των Κοινοτήτων. Ε, δεν θα πρέπει να γελιόμαστε. Παίζουμε ε, κορώνα γράμματα το μέλλον των επόμενων γενναιών. Δεν θα πρέπει άλλο να χρονοτριβούμε. Ο κύριο Συναδίνο, για ένα λεπτό. Οι αποφάσει για τι κατεφημισμών ελεύθερε και δίκαιε εκλογέ δεν εξυπηρετούν τη δημοκρατία, αλλά αντιθέτω την αδιαφάνεια και την κομματοκρατία. Δημιουργούνται ανύπαρκτοι εχθροί, ώστε οι ευρωπαϊκέ ελίτ να μην αντιμετωπίσουν την αλλαγή και τα λάθη που οι ίδιε διέπραξαν. Η απάντηση σαφή. Μόνο πατριωτικά κινήματα μπορούν να αποφέρουν μια υπεύθυνη διακυβέρνηση εποφελία των εντολέων πολιτών και την επιστροφή στη συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων κυρίαρχων κρατών. επιπλέον επισημαίνω πω ενώ καταδικάζεται την παραπληροφόρηση η ευρωπαϊκή ένωση επιδιώκει ανοιχτά την προώθηση πολιτικών ιδεών και την καλλιέργεια συγκεκριμένη νοοτροπία και αντιλήψεων όπω και οι πληρωμένοι πράκτορε τη τουρκική μυτ παραπληροφορούν αλωνίζοντα ανενόχλητοι μέσα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο όπω οι αλβανοί δίθεν τσάμιδε πω γνήσιοι δοσύλλογοι εξυπηρετούν το ιδεολόγημα τη μεγάλη αλβανία όπω όσοι πολιτικοί προδότε παρέδωσαν το όνομα της μακεδονίας στους σλαβοαλβανούς σκοπιανούς παραχαράσσοντας την ιστορία και παραπεραιώντας την αλήθεια. σε αυτά η ευρώπη δεν είναι θεατής αλλά συμμέτοχη εναντίον της ασφάλειας και των ζωτικών συμφερόντων των κρατών μελών όπως η ελλάδα. προφανώς η απειλή βρίσκεται εντός των τυχών. γι' αυτό το ηνωμένο βασίλειο καλώς αποχωρεί και καλώς ο σαλβίνη σας γυρίζει την πλάτη. ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν θέλει να ε, τιμωρήσει τους ε, Βρετανούς, κανείς δεν θέλει να τους ε, ταπεινώσει. Εμείς τους θέλουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα ήταν πολύ καλοί εταίροι. Αλλά το να χρησιμοποιείτε αυτό το επιχείρημα ότι θέλουμε να τους ταπεινώσουμε, αυτό αποδεικνύει ότι οι υπέρμαχοι του Brexit δεν έχουν κανένα άλλο επιχείρημα παρά χρησιμοποιούν αυτό το τετριμένο περί τιμωρίας. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να καταλήξει σε μία απόφαση. Το Λονδίνο πρέπει να μιλήσει στο εσωτερικό του, μεταξύ τους να βρουν μια λύση. Αυτός είναι ο δρόμος, είναι ο δρόμος για να δοθεί καλύτερη λύση, καλύτερο μέλλον στο Βρετανικό λαό. Ως εκ τούτου είναι απολύτως απαραίτητο ε, να ληφθεί μια απόφαση, όπως το πρότεινε και το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, ή να έχουμε μια μακρύτερη παράταση με βάση την ε, συμφωνία που έχει μέχρι τώρα επιτευχθεί. Αν όμως ένα κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να αποφασίσει, τότε το κοινοβούλιο να μεταθέσει την απόφαση στο λαό με νέες εκλογές ή με ένα νέο δημοψήφισμα. Αυτή είναι πεπατημένη στη δημοκρατία. Ένα λεπτό, η κυρία Ζίπελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ στις 19 ε, Μαρτίου στην Ουταλία ε, κατασχέθηκε η Μάρε Γιούνιο και πολλοί θεωρούν ότι θα πρέπει να καταδικαστούν υπεύθυνοι μέχρι και 20 χρόνια. Στο Συμβούλιο όμως δεν ελέγχθη τίποτα. Ούτε ελέγχθηκε τίποτα για όλα αυτά τα καθημερινά βασανιστήρια και τους βιασμούς, επίσης τους, τα υποτιθέμενα στους υποτιθέμενους επίσημους καταβλισμούς της Λιβύης. Όμως εμείς δεν θα σιωπάσουμε όταν κράτη-μέλη καταπατούν τα χριστιανικά δικαιώματα και απεκδίονται των ευθυνών τους. Ε, κύριε Τούσκ, ε, ο κύριος Τούσκ νομίζω δεν μας ακούει, αλλά ξέρετε τι κάνετε, εσείς τιμωρείτε τους διασώστες. Επιτέλους, ε, άρετε το μπλοκάρισμα στο Λονδίνο, να γκρίνεται για τη νέα συμφωνία του Δοβλίνου, όπως την έχουμε αποφασίσει, γιατί δεν πρέπει να τιμωρείται η διάσωση των πολιτών, αλλά το να αρνείται κανείς τη βοήθεια σε ανθρώπους που κινδυνεύουν, αυτό θα πρέπει να τιμωρείται. Η κυρία Χιούπνερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Για 120 μέρες ήταν επιτάπητος η Συμφωνία Αποχώρησης και πάλι σήμερα είναι κρίσιμη εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ε, θα είναι καθοριστικά τα αποτελέσματα για τους πολίτες. Τα όρια της αβεβαιότητας, οικονομικής και πολιτικής, φτάνουν στα άκρα κατά τον Brexit. Δεν ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη έκαναν όλες τις προσπάθειες για να είναι ε, σίγουρη αυτή η διαδικασία. Η απόφαση της Πέμπτης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δίνει ακόμα μια ασφάλεια δικαίου, όχι μόνο στην ε, Συμφωνία Αποχώρησης, αλλά σε όλη τη διαδικασία. Τέλος, αν η επιλογή για μακρότερη παράταση συζητηθεί σοβαρά, αν στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνει μια διαπαραταξιακή συζήτηση και απόφαση για νέα πολιτική δήλωση, ε, καλούμε τα βρετανικά πολιτικά κόμματα να ε, το κάνουν με τρόπο που θα σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών και θα αποφεύγει τη δημιουργία βεβαιότητας ανάμεσά τους. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό ο κύριος Λάινεν. Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής ε, πολύ σωστά δεν ασχολήθηκε μόνο με τον Brexit, αλλά βλέπουμε από τη συζήτηση αυτή πώς η ενεργεία μας στοιχίζει αυτό το θέμα, στερώντας την από άλλα θέματα σημαντικά, όπως ε, αλλαγή κλίματος και Κίνα. Αυτά πάνε μαζί. Είναι εταίρος η Κίνα στην ε, προστασία του κλίματος, αλλά είναι αντίπαλος στις τεχνολογίες. Έχει στρατηγική σαφή για την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών προχωρούν τάχιστα στις κυψέλες, στις μπαταρίες αυτοκινήτου. Εμείς έχουμε βιομηχανική πολιτική για το κλίμα, για τις σχετικές τεχνολογίες αποθήκευσης, παραγωγής μπαταριών αυτοκινήτων, για την βιομηχανία χάλιβα, την τσιμεντοβιομηχανία. Πρέπει να δουλέψουμε εκεί και η Κίνα είναι τέρος αλλά είναι και ένας συστημικός ανταγωνιστής και αυτά θα πρέπει να τα δούμε κατά τη σύνοδο. Πρέπει να προστατευτούμε χωρίς να είμαστε προστατευτικοί, χωρίς προστατευτισμό. Ο κύριος Κέλλη, ένα λεπτό. Εγώ συνοψίζω τον Brexit ως εξή. Το Brexit μας τρελαίνει. Όλα είναι πολύ άσχημα σχετικά με αυτό. Αυτά τα πισωγυρίσματα ε, δημιουργούν ε, ε, αβεβαιότητα. Ελπίζομαι ότι κάποια στιγμή τα πνεύματα θα συναντηθούν στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ε, και θα ληφθούν υπόψη οι διαδηλώσεις της, ε, του τελευταίου Σαββατοκύριακου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τις αναφορές που υπεγράφησαν. Ελπίζω να πάρει αποφασιστική απόφαση το Κοινοβούλιο για να ε, αποφευχθεί το no deal θα επιφέρει μεγάλη καταστροφή. Ε, μπορούμε να έχουμε παράταση, αλλά αν δεν ληφθεί απόφαση, τότε ε, όλοι θα συνεχίσουν να ανησυχούν. Ε, ε, ο κόσμος εξακολουθεί να απορεί για τη συνέχεια που θα δοθεί, αλλά οι υπέρμαχοι του Brexit δεν έχουν ιδέα για να τον καθοδηγήσουν. βλέπω ότι ορισμένοι το είδαν αυτό πολύ, την ομιλία σας πολύ διασκεδαστική. Ευχαριστώ Σον. Ε, ο κ. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αξιοπερίεργο ότι κανένα μέλος του κυβερνώντος κόμματος της Βρετανίας δεν ήρθε να μιλήσει. Γιατί τρομοκρατούνται από, το, από αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Και ε, μόνο ο κύριος Φάρατς βέβαια βρίσκεται εδώ από τους Βρετανούς. φοβούνται γιατί έδωσαν υποσχέσεις ότι θα είναι ένα πράγμα το Brexit και αποδεικνύεται ότι είναι τελείως διαφορετικό. Ε, όπως ε, ε, πολλοί πολιτικοί που δίνουν υποσχέσεις και μετά εξαφανίζονται και πάνε αλλού με τα τζέτ τους. Εσείς είστε υπεύθυνοι για την εθνική ταπείνωση και κανένας άλλος. Μην κατηγορείτε άλλους. Και ήρθε η ώρα να αναλάβετε την ευθύνη των ψεμάτων και της υποκρισίας σας η οποία γονάτισε τη χώρα. Κύριε Τούς, και ευχαριστώ για το μήνυμα αλληλεγγύης, το δεχόμαστε με σεβασμό. Υπάρχει μεγάλο κίνημα στη Βρετανία υπέρ της παραμονής. Δεν θα φύγουμε. Θέλουμε να νικήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και είμαστε περήφανοι που σας έχουμε μαζί μας. Και ένα διαδικαστικό, κύριε Αντιπρόεδρε. Ο κύριος Μπάτεν μίλησε για κουίσλινγκ και για προδότες. Τέτοιου είδους γλώσσα είναι εντελώς απαράδεκτη σε αυτό το κοινοβούλιο και σε οποιοδήποτε κοινοβούλιο και οπουδήποτε. Και θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. and the House supports you. Φαίνεται ότι η Ομίγυρη συμφωνεί μαζί σας. Ο κύριος Ρανζέλ, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε Τούσκ, αγαπητέ επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, Μισελ Μπαρνιέ, το πρώτο σημείο που θα ήθελα να διευκρινίσω ε, για την Βρετανική Βουλή, ε, κύριε Φάρετς, το είπατε ήδη, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλόπιστη, καλοπροαίρετη και απέναντι στον Βρετανικό λαό και απέναντι στους διαπραγματευτές της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσω είναι το θέμα του Brexit. Δεν είναι μόνο ένα θέμα προσδιορισμού μιας διαπραγμάτευσης και κάποιων δικαιωμάτων. να δούμε τι δικαιώματα έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Βρετανοί πολίτες, όπου και αν βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ταυτόχρονα θα πρέπει να στηρίξουμε και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Αυτό όμω λείπει προς το παρόν. Γιατί υπάρχει μια βεβαιότητα, δημιουργείται μια αποσταθεροποίηση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με αυτές τις παρατάσεις. Το είδα αυτό με τους ε, ε, Πορτογάλους εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου ε, και μου έχουν πει πολλοί και στην Πορτογαλία ότι ανεξάρτητα από τις ε, συμφωνίες που έχουμε για το θεωρητικό θεσμικό πλαίσιο, αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από την αβεβαιότητα και την αστάθεια που υπάρχει, γιατί δεν είναι προβλέψιμο το μέλλον ούτε των πολιτών ούτε των επιχειρήσεων. Ο κύριος Σίλβα Περέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Συμβούλιο έλαβε καλές αποφάσεις ε, για την πολύ σύντομη παράταση του Brexit και του άρθρου 50. Κάτι που είναι ε, επιτρεπτό μέχρι τις 22 Μαΐου και εφόσον φυσικά ε, η Βουλή των Κοινοτήτων εγκρίνει τη συμφωνία για την αποχώρηση. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το πολύ μέχρι τις 12 Απριλίου για να διευκρινίσει άπαξη διαπαντός στις προθέσεις του. Και υπάρχει εύλογος λόγος για κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχθεί ε, αυτή αυτό το πρόβλημα του Brexit, αυτή η γκάφα του Brexit να μολύνει τις ευρωεκλογέ και να προκαλέσει ένα δικαστικό πόλεμο και κρίση ε, νομιμοποίησης για τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως συγητής ε, της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιέλαβα μία ρήτρα που λέει ότι η ε, νέα σύνδεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ισχύσει μετά την υλοποίηση του Brexit. Αν δεν εγκριθεί συμφωνία και δεν αποτραπεί η περίπτωση του no deal, η μόνη παράταση του άρθρου 50 ε, που θα ήταν αποδεκτή θα είναι μια πιο μακροπρόθεσμη παράταση που θα επιτρέψει Βρετανούς πολίτες να λάβουν μέρος σε ευρωεκλογέ και να έχει χρόνο και το Ηνωμένο Βασίλειο να χαράξει τη νέα στρατηγική του για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής ε, στον κατάλογο μου, αλλά όχι λιγότερο εκλεκτός από τους υπόλοιπους, είναι ο κύριο Άσχορθ και δεν θα σας δώσω επιπλέον χρόνο γιατί δεν είναι η τελευταία σας ομιλία, αλλιώς θα σας έδινα και λίγο παραπάνω χρόνο. Κύριε Τούσκ, κύριε Πρόεδρε Τούσκ, εκ μέρου ε, του εκατομμυρίου των ανθρώπων που κατέβηκαν στους δρόμους στο Λονδίνο, εκ μέρου των 6 εκατομμυρίων ανθρώπων που υπέγραψαν ε, το αίτημα και εκ μέρου του 63% των Βρετανών οι οποίοι δεν υπερψήφισαν το Brexit, θέλω να σας πω, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή σας και σας διαβεβαιώνω ότι ο κύριος Φαράτζ δεν ομιλεί εξ ονόματος του 63% των πολιτών. Και θα ήθελα να προσθέσω και ένα άλλο σχόλιο προς τους Ευρωπαίους ότι για πάνω από 25 χρόνια ε, κανένας Βρετανός Πρωθυπουργό δεν εξήγησε στους Βρετανούς το τι ακριβώς έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα ωφέλη που προσφέρει και γιατί παίζει ρόλο αυτό. Ε, ποτέ κανείς δεν υπερασπίστηκε και δεν ε, διέψευσε αναλήθειες και ποτέ κανείς δεν εξήγησε αποφάσεις του Συμβουλίου. Γι' αυτό το λόγο ο Βρετανικός του τύπος μετά από μια εκστρατεία 20 ετών των λαϊκιστών ε, βασισμένη εκστρατεία σε αναλήθειες, ψέματα και απάτες ε, οδήγησε σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Η Βρετανία είναι λυπημένη. Είναι ένας διχασμένος λαός, όπως ποτέ στο παρελθόν. Ε, το Βρετανικό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε κρίση. Γι' αυτό λοιπόν το Brexit ας είναι ε, ένα ε, κάτι, μια προειδοποίηση για τους Ευρωπαίους πολίτες, στους οποίους θέλω να πω το εξής. Εσείς είσαστε η γενιά που ζήσατε την μακρύτερη περίοδο ειρήνης και το καλύτερο επίπεδο διαβίωσης που υπήρξε ποτέ. Ποτέ λοιπόν, ποτέ να μην το θεωρείτε αυτό δεδομένο. Να το εκτιμάτε, να αγωνίζεστε γι' αυτό και να το υπερασπίζεστε κάθε ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Άσουερθ. Ε, ήταν σωστή η απόφασή μου να σας δώσω το λόγο και ε, μας προειδοποιήσατε αποτελεσματικά γιατί μιλήσατε ε, με ενθουσιασμό για τη χώρα σας. Η κυρία Σιόντροβα. Ένα λεπτό το πόλι και δώστε το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το να παίρνει κανείς το λόγο μετά τον κύριο Άσχορτ ε, δεν του διευκολύνει τα πράγματα. Ε, σέβομαι απόλυτα αυτά που είπατε και πιστεύω ότι κάθε Βρετανός θα πρέπει να ακούσει αυτά που είπε ο κύριος Άσχορτ και όχι αυτά που είπε ο κύριος Λεγκούτκο. Γιατί μίλησε και αποτροπή ο κύριος Λεγκούτκο, σαν να μην έχει την ευκαιρία να ε, ψηφίσει το κοινοβούλιο μια αξιοπρεπή συμφωνία και ένα αξιοπρεπές ε, Brexit. Οι Βρετανοί αποφασίζουν για το μέλλον τους, όχι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι για αυτούς. Ευχαριστώ κύριε Τούς και ευχαριστώ που μας εξηγήσατε τις προετοιμασίες που κάνετε για τη Σύνοδο Κορυφής με την Κίνα. Μας μιλήσατε επίσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης θα πρέπει να είναι τμήμα οποιασδήποτε εμπορική συμφωνίας. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει σε πολλές εκθέσεις του τη σημασία που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να το λάβουν υπόψη και ισχύει και για μας το ίδιο. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε ο κύριος Εμμανουέλ Μακρό με τις προτάσεις του. Ο κύριο Λόπε Αγγιλάρ, προσπαθώ να ικανοποιήσω όλου του συναδέλφου που ζήτησαν το λόγο στο ΚΑΤΣΔΙΑ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του ΣΚΠΟΛΗ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένω ήμασταν επικριτικοί απέναντι στο Συμβούλιο. Όχι όμω και αυτή τη φορά. Κάνετε το σωστό με πολύ σωστή ημερομηνία. Όχι άλλη παράταση. 12 Απριλίου για να βρει η Βρετανική Βουλή μία διέξοδο, ένα σχέδιο για το Brexit όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από το λαβύρινθο στον οποίο έχουν εγκλωβιστεί και δεν βρίσκουν τη διέξοδο. Έχουμε συμπάθεια προς τα εκατομμύρια των Βρετανών που έχουν κατεβεί στους δρόμους. Αλλά δεν θα πρέπει να ε, δείξουμε υπομονή απέναντι στους ανεύθυνους δημαγωγούς και δημοκόπους που έκαναν μεγάλη ζημία προς το Βρετανικό λαό με τη χειραγώγηση που εφάρμοσαν. Θα πρέπει επίση να πούμε τώρα ρητά και κατηγορηματικά ότι τώρα είναι η στιγμή. Είναι και είναι η ώρα. Άλλη παράταση δεν επιτρέπεται. Το κακό μαντάτο είναι ότι δεν μα άφησαν ουσιαστικά να μιλήσουμε για τίποτα άλλο. Η χαρμόσυνη πάντω είδηση είναι ότι ήδη η κλεψίδρα έχει αρχίσει και τρέχει. Θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα στην Βουλή των Κοινοτήτων να διευκρινίσουν τη θέση τους ή έξοδος ή ανάκληση του άρθρου 50. Και αν ναι, θα πρέπει να γίνουν ευρωεκλογέ αν θέλουν περισσότερη ε, παράταση. Η κυρία Τόμασιτς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Brexit ε, ε, είναι μια χαοτική διαδικασία. Ε, πριν από τρία χρόνια αποφάσισαν οι Βρετανοί για την έξοδο και ακόμη δεν είναι σίγουρο αν θέλουν να την υλοποιήσουν πότε και υπό ποιου όρου. Αυτό είναι ντροπή. Όχι μόνο για τη Βρετανική κυβέρνηση που ήταν ανίκανη να υλοποιήσει τι προσδοκίε των πολιτών τη, αλλά και για την Ευρώπη που η Ένωση Εθνών δεν σημαίνει τίποτα. Και πριν ε, το Brexit ε, το κατεστημένο γνωούσε την βούληση του πολίτη. Και αυτό φάνηκε στα πολλά μαθήματα που όμως ε, δεν, στα πολλά παθήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έγιναν μαθήματα όμως δεν είχε μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο πρόβλημα με τον Brexit. Τι, να πούμε με άλλες πιο μικρές χώρες που δεν είναι νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δέχτηκαν, αναγκάστηκαν να δεχτούν το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Θα πρέπει λοιπόν όλα να τα λάβουμε υπόψη. Γιατί όταν έρχεται η ώρα να πληρώσουμε το λογαριασμό, δεν θα πρέπει να αφήνουμε τον άλλον να πληρώνει τα σπασμένα. Ευχαριστώ. Κυρία Φάουτμανς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι κάναμε καλή συζήτηση. Θα ήθελα να ε, σας πω κάτι εδώ και καιρό κύριε Φάρατζ. Σταματήστε να ψεύδεστε. Ακόμα και σήμερα εξακολουθείτε να ψεύδεστε. Και στον κύριο Άσουορθ ε, κάτι. Νομίζω ότι στείλατε το σωστό μήνυμα. Νομίζω ότι πρέπει να παλέψουμε για την Ευρώπη. Πρέπει να ανανεώσουμε την Ευρώπη. Αυτό είναι το δίδαγμα για όλους μας ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θέλω αυτό να κάνουμε στην προεκλογική εκστρατεία. Να δώσουμε μάχη για την Ευρώπη, να την προστατέψουμε για να γνωρίζουμε τι κάνει η Ευρώπη για μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φερκόνεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Brexit είναι μεγάλη τραγωδία και δείχνει πού οδηγεί ο λαϊκισμός. Ε, πρόκειται για γόρδιο δεσμό στο Ηνωμένο Βασίλειο που επηρεάζει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να βοηθήσει βρίσκοντας λύση, γιατί η κατάσταση είναι δυσχερέστατη. Το Brexit έδειξε ε, τι μπορεί ε, να ε, συμβεί σε έναν λαό που έχει παρασύρθει και χάνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελεύθερη διακίνηση μεταξύ άλλων. Ε, ε, πρέπει να είναι σαφές ε, σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες τι μπορεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υποστηρίξουμε μια διαδικασία όπου θα βρει μια διαρκή λύση το Ηνωμένο Βασίλειο και γι' αυτό το πιο ρεαλιστικό θα ήταν ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Ο κύριος Καπούτο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα μιλήσω για το Brexit, θα μιλήσω για το κλίμα. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι διαμαρτύρονται σε ολόκληρο τον κόσμο για το μέλλον του ε, και αυτό το στήριξε η Ολομέλειά μα. Αλλά δυστυχώ δεν το έλαβε υπόψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σίγουρα είναι απαραίτητο να γίνουν περισσότερε προσπάθειε σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπιστεί το κλίμα, αλλά πέρα από τα προγράμματα, η συνάντηση κορφή δεν κατόρθωσε να δώσει μια σαφή γραμμή για το θέμα της μη χρήση άνθρακα. Ε, το, ο στόχος δεν αναφέρεται καθόλου, απλά η που απάγεται στα βιομηχανικά συμφέροντα και αυτά αποκρύπτουν την πραγματικότητα ότι θα πρέπει κάθε χώρα να είναι σε θέση να διαλέξει το δικό του το ενεργειακό μείγμα και σε ορισμένε περιπτώσεις να διαφυλάξει τη χρήση των ε, ορυκτών καυσιμών που όμως αυτά βλάπτουν το κλίμα και την οικονομία το σπίτι μας ε, καίγεται, αλλά εμείς ε, εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε ότι ε, το πρόβλημα οφείλεται κάπου αλλού. Η κυρία Γουκασεύσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ουδής στην αίθουσα δεν πιστεύει ότι οι Βρετανοί θα λάβουν απόφαση για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το πιστέψαμε ε, είδαμε από την ιστορία ότι πολλές φορές οι πολίτες ενδίδουν στο λαϊκισμό και ε, ανέδωσαν στα σχόλια που εκφώνησαν άνθρωποι όπως ο κύριος Φαράζ. Σήμερα έχουμε ε, χάος, χαοτική κατάσταση και ζημίες που υφίσταται η Βρετανική οικονομία λόγω αυτής της απόφασης. Πάντως έχω την ελπίδα ότι το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, το παράδειγμα του Brexit και της χαοτικής κατάστασης που προκάλεσε θα είναι καλό μάθημα για όλους εκείνους στην Ευρώπη που ονειρεύονται την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ε, θα λαχταρούσαν να... Ε, τονίσουν το μίσος τους κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην έχουμε λαϊκιστές να μην έχουμε ανθρώπους που πολύ ευχαρίστω δέχονται τα κονδύλια και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παρόλα αυτά την απεχθάνονται και θέλουν να αποχωρήσουν από αυτή το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ κύριο Σπυρίνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην αρχή αυτής της ε, συνεδρίασης, ο πρόεδρος Τούσκ ε, ανέφερε ένα κείμενο στα από τα συμπεράσματα η ισχυρή οικονομική βάση είναι κέρια σημασίας για την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Και υπογράμμισε, κυρία, κυρία Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να υποβάλει μέχρι το τέλος του 2019 ένα μακρό προόραμα για τη βιομηχανία της Ευρώπης με συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή του. Κύριε Πρόεδρε, απευθύνω έκκληση σε εσά και μέσω ημών στον πρόεδρο Τούσκο που έφυγε αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπω ότι επιστρέφει και προς τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν. Σκεφτείτε προσεκτικά τι σημαίνει η διατύπωση αυτή. Μέχρι το τέλος του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα μακρόπνο όραμα. Αυτό δεν μπορεί να είναι τεχνοκρατικό εγχείρημα, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να λάβει υπόψη την αποβιομηχάνηση της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στις προηγούμενες δεκαετίες. Αν θέλουμε ισορροπημένη βιομηχανία στο μέλλον, πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτή την κεντρική πρόκληση για τη βιομηχανία, τις θέσεις και την ανάπτυξη. Στην αρχή της συνεδρίασης, κυρία Πρόεδρε, έπρεπε να χειριστείτε το θέμα της κινητικότητας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα υπηρεσιών από την Ανατολική Ευρώπη που εκδιώκεται από την αγορά χρησιμοποιώντας ε, θεμη ανησυχίες κοινωνικές και εργασιακές. Πρέπει να ε, δράσω με πάση θυσία. Θα πρέπει προσωπικά να παρακολουθήσετε πώς αυτό το κείμενο για το βιομηχανικό μέλλον θα μεταφερθεί από το ένα κοινοβούλιο στο άλλο, από τη μία επιτροπή στην άλλη, διότι αυτό είναι κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου επιτρέψατε λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Σαρμπάτη. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τη συζήτηση. Ε, νομίζω ότι εδώ, σε αυτό το σπίτι, έχουμε πολλούς φαρισαίους. Μάλιστα, είναι και μερικοί που είναι φανατικοί φαρισαίοι. Πολλοί μιλάνε για τους Βρετανούς, αλλά στη τελική ανάλυση αυτό το σπίτι και αυτό το συμβούλιο τους έδιωξε. Για την ε, Ελλάδα ξεπεράστηκε κάθε κόκκινη γραμμή που μπορούσε να φανταστεί κανείς για να μείνουν αυτοί στην Ευρωζώνη. Και στον Κάμερον του απαγορέψαμε να συζητήσει την αρχή της ελεύθερης δεύτερης μετακίνησης. Εάν λοιπόν αυτό το είχαμε συζητήσει και είχαμε δώσει μια απάντηση στον Κάμερον, τότε και το Brexit ε, θα ήταν τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα. Η ελεύθερη μετακίνηση, η κινητικότητα ήταν εκείνη που οδήγησε τους Βρετανούς να υπερψηφίσουν υπέρ του Brexit. Ακούγοντας αυτά τα φαρισαϊκά και σε εσά απευθύνομαι κύριε Μπούλμαν με τις αιτιάσεις σας ε, και ο κύριος Φερχόφτσατ και εσείς γιατί δεν μπορεί πια κανείς ε, να το αντέξει πώς έχουν καβαλήσει το καλάμι οι άνθρωποι αυτοί και τρέχουν ασυγκράτητοι. Το αποτέλεσμα στη Μεγάλη Βρετανία είναι ότι πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα συμμετοχή δεύτερη κατηγορία ή στο Brexit και σύγκρουση με την Ιρλανδία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν υπήρχε το πρόβλημα με την Ιρλανδία θα υπήρχε κάποια λύση. Αλλά υπάρχει ένα δίλημα από το οποίο δεν μπορεί κανεί να βγει. Οι Βρετανοί ποτέ δεν θα θελήσουν να είναι μέλο δεύτερη κατηγορία, να μην μπορούν να συναποφασίσουν, να πληρώνουν και να να μην έχουν ε, τη δυνατότητα να συνάψουν ελεύθερες ελεύθερα εμπορικές συμφωνίε. Γι' αυτό λοιπόν είναι σωστό να ξαναγίνει δημοψήφισμα και στην περίπτωση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να πούν στου Βρετανού. εντάξει, δεχόμαστε του όρου σα. συζητάμε του όρου σα. Κυρία Πρόεδρε, αφήσατε κάποιον να μιλήσει δύο λεπτά και εγώ επιτρέψτε μου να πω μία τελευταία πρόταση. Πρέπει να πούμε στου Βρετανού ότι είναι ευπρόσδεκτο να τους πούμε ότι έχουν το δικαίωμα αυτά που τους αφορούν να τα ρυθμίσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχαριστημένοι. Και αν τα κάνουμε όλα αυτά θα επανέλθουν. Ο κύριος Επιτίδιος παρακαλώ. Ε, grazie, Presidente. Ο τρόπος με τον οποίο ε, χειρίζεται το θέμα του Brexit η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενδεικτικός της εσφαλμένης πολιτικής που εφαρμόζει για την αντιμετώπιση και όλων των σοβαρών θεμάτων που έχει να αντιμετωπίσει. αντί να αναλογιστεί και να προσπαθήσει να διορθώσει τα λάθη τα οποία διέπραξαν και υποχρέωσαν το βρετανικό λαό να επιδιώξει την έξοδό του από την ευρωπαϊκή ένωση επιθυμεί να τιμωρήσει και να εξευτελίσει τον βρετανικό λαό. με το ίδιο πνεύμα με την ίδια φιλοσοφία επιδιώκει να τιμωρήσει την ουγγαρία την πολωνία με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 εναντίον τους το κόμμα φιντές του κυρίου όρμπαν και επίσης με αυτό το πνεύμα επί εννέα συνεχή χρόνια τιμωρεί την ελλάδα και τον ελληνικό λαό τον οποίο έχει εξαθλιώσει με τα συνεχή μνημόνια που του έχει επιβάλει και δεν επιθυμεί να μειώσει το επαχθές χρέος το οποίο έχει υποστεί ο ελληνικός λαός. τιμωρία λοιπόν και μόνο τιμωρία αυτή είναι η φιλοσοφία της ευρωπαϊκής Ενώσεω και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μετά από δύο μήνες θα εμφανιστεί σε αυτό το ευρωκοινοβούλιο η αρχαία θεά της τιμωρίας η νέμεσης υπό την παρουσία πολλών πατριωτικών κομμάτων στον χώρο αυτό. Ευχαριστώ. Όπω Σπυράκη, παρακαλώ. Πρόεδρε, όπως ξέρετε και από τη μητέρα σας, οι αρχαίοι Έλληνε έλεγαν «ουδέν κακόν, αμυγές καλού» τι συμβαίνει λοιπόν με το χάος που πάει να δημιουργηθεί από το brexit; μπορούμε να δούμε μέσα από εκεί ότι αποκαλύπτονται οι επιπτώσεις του λαϊκισμού τα απόλυτα ψέματα που σέρβιρε ο κύριος ή οι απόλυτες ψευδεστήσει που σέρβιραν οι ομοειδεάτες του. τι συμβαίνει λοιπόν μέσα από το χάος του brexit; βλέπουμε τον κίνδυνο να συμπεριφερθούμε τιμωρητικά απέναντι στους πολίτες του ηνωμένου βασιλείου και δεν πρέπει να το κάνουμε. πρέπει να τους δώσουμε όλες τις ευκαιρίες να επιλέξουν. τι συμβαίνει μέσα από το χάος του brexit; βλέπουμε τον κίνδυνο να πληγώσουμε και εμείς τους εαυτούς μας με μια άτακτη κίνηση με μια ασύντακτη κίνηση brexit. τι νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε; να δείξουμε πως είμαστε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να δώσουμε στους πολίτες του ηνωμένου βασιλείου την ευκαιρία να συμπεριφερθούν με νυφαλιότητα να κρίνουν και να αποφασίσουν ξανά για το δικό τους μέλλον να στηρίξουμε ένα δεύτερο δημοψήφισμα. σας ευχαριστώ πολύ ο Κύριε Πρόεδρε, ο κύριο Βέμπερ μίλησε για το άρθρο 7 τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα ήθελε να με επικρατεί δηλαδή και να κυριαρχεί στις χώρες και στις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να το παρακάμψουμε αυτό το άρθρο. Δηλαδή, με τα αποτελέσματα αυτά, όχι αυτά που προβλέπει η συνθήκη, αλλά αυτά που θα ήθελε ο κύριος ε, Βέμπερο, κατά πάσα πιθανότητα μελλοντικό πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έτσι να το ερμηνεύσουμε, όπως εκείνος θέλει. Αλλά τι γίνεται με τη θέση των χωρών που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλειοψηφία που θα ήθελε να συνεχίσει αυτή την περιπέτεια εις βάρος της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, ίσως θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη ότι η συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε να ληφθούν τόσο εύκολε αποφάσει για να διχάζουν την Ευρώπη. Τώρα, αν για τον κύριο Βέμπερ δεν, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο πλουραλισμός στα κράτη-μέλη, το κράτος δικαίου, τα ελάχιστα, τα θεμελιώδη δικαιώματα των μειονοτήτων και τα, το δικαίωμα της μειοψηφία να έχει διαφορετική γνώμη, τέτοια Ευρώπη θέλετε, αυτή την Ευρώπη προασπίζετε. Γιατί έτσι θα εμβαθύνετε κάποιες διαιρέσεις και διχασμούς που ήδη είναι πολύ άριθμοι. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο Μισελ Μπαρνιέ, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Πολύ σημαντική η συζήτηση, κατά την οποία ακούσαμε τον Πρόεδρο Ιούνκερ και ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν και εγώ σας ε, ακούσαμε με ιδιαίτερη προσοχή και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Άκουσα την πρόσκληση του Προέδρου Ντόναλτ Τούσκ, τον οποίο ευχαριστώ και προσωπικά που έλαβε μέρος ε, στις συζητήσεις ε, του Συμβουλίου, τα αποτελέσματα των οποίων μας παρουσίασε σήμερα το πρωί. Αυτή η διαπραγμάτευση για τον Brexit είναι όντως έκτακτη, είναι εξαιρετική και είναι έκτακτη και από άποψη σοβαρότητας και από άποψη ευθύνης. Ευθύνης που βαρύνει όλους τους ε, ηγέτες, όλους τους αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Θα πρέπει με πολύ σοβαρό, υπεύθυνο και αντικειμενικό τρόπο να λεφθούν οι αποφάσει όπως γίνεται και στι διαπραγματεύσει. Πριν από δύο χρόνια, ο πρόεδρο Γιουνκέρ και ο πρόεδρο Τούσκ με την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μου ενέθεσαν αυτή την αποστολή τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Και εδώ και μία διετία, κυρίε και κύριοι, εδώ και μία διετία και εγώ, όπως και εσείς, γιατί ε, αυτό το σημείο το επισήμενο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ε, Ευρωπαίων πολιτών κατά προτεραιότητα. Όπως είπαν και ο κύριος Φεχόφστατ, ο κύριος Βέμπερ, ο κύριος Γουαλτιέρη, ο κύριος Μπούλβαν, η Γκάμπι Τσίμερ και άλλοι. Αυτό ήταν η προτεραιότητα μας, η διασφάλιση των 4,5 εκατομμυρίων πολιτών 3,5 ε, εκατομμύρια ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο που συμμετέχουν στην οικονομία της χώρας. 1,5 εκατομμύριο Ευρω... Βρετανοί πολίτες διαβίουν και εργάζονται στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτή η διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών των πολιτών, όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα ύψη την προτεραιότητά μας. Και ευελπιστώντας ότι θα ληφθεί μια συμφωνία, ακόμη και αν προετοιμαστούμε και έχουμε προετοιμαστεί για μια έλλειψη συμφωνία. αυτή η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους θα εξακολουθεί να είναι η υψηλή προτεραιότητά μα. Εδώ και δύο χρόνια εργαζόμαστε και εγώ και το επιτελείο μου, με τον ίδιο και αμύωτο σεβασμό προ το Ηνωμένο Βασίλειο. Τρέφουμε ιδιαίτερο θαυμασμό και προ το Ηνωμένο Βασίλειο. Το έχω πει θαυμασμό για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για τον μεγάλο αριθμό των ηγετών άνδρων και γυναικών που έχει στην ιστορία, χωρίς να ξεχνούμε την αλληλεγγύη που έδειξε το Ηνωμένο Βασίλειο στις ε, πιο σημαντικές στιγμές του 20ου αιώνα απέναντι προς εμάς. Και αυτός ο σεβασμός διέπει τις εργασίες μας. Και αυτός ο σεβασμός, κύριε και της κυρίαρχης απόφασης των ε, Βρετανών πολιτών, της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών. Σεβόμαστε αυτή την απόφαση. Ακόμη και μας θλίβει, παρόλα αυτά τη σεβόμαστε και προσπαθούμε να την υλοποιήσουμε συνειδητά, μεθοδικά, εδώ και μία διετία. Αυτό κάνουμε κύριε Φαράς. Ούτε ένας άνθρωπος στις Βρυξέλλες δεν προσπαθεί να κλέψει τον Brexit ή να εκτρέψει την ετοιμιγορία των Βρετανοπολιτών. Δεν έκανα η Βρυξέλλες αυτή την επιλογή. Εσείς κάνατε την επιλογή να εξέλθετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποχωρήσετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς λοιπόν θα πρέπει να επομιστείτε τις ευθύνες σας απέναντι στις συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης και κανείς άλλος. Εδώ και δύο χρόνια και με αυτό το σεβασμό που διαπνέει τις διαπραγματεύσεις προσπαθούμε να υλοποιήσουμε την απόφαση αυτή. Ο κύριος Λεγκούτκο έφυγε και δεν θα με ακούσει. Αλλά σα διαβεβαιώ ότι ούτε μία στιγμή, ούτε ένα δευτερόλεπτο κατά τη διετία αυτή δεν είχαμε στην συμπεριφορά μας οποιαδήποτε ένδειξη ρεβανσισμού, εκδίκησης ή ε, επιθυμίας ταπείνωσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ούτε μία στιγμή δεν πέρασε κάτι τέτοιο από το μυαλό μας ή δεν δείξαμε κάτι τέτοιο με τη συμπεριφορά μας. Πριν από λίγο, η πρόεδρος Μαγκίνες το δήλωσε, αλλά και ο κύριος Ονκέλη και ο κύριος Νίκολσον. Ακούμε ιδιαίτερη προσοχή τα σχόλιά σας και την κυρία Άντερσον και την κυρία Ντότζ. Εδώ και μία διετία προσπαθούμε υπομονετικά να βρούμε λύσεις λειτουργικές για το σοβαρότερο πρόβλημα που δημιούργησε το Brexit και που βρίσκεται φυσικά στην Ιρλανδία. Το σοβαρότερο πρόβλημα κίνδυνος για τη σταθερότητα και την ειρήνη στο νησί, στην οποία συμμετείχαμε από εδώ και μία ε, εδώ και πολλά χρόνια με τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, τη συμφωνία του Belfast. Και λίγα λόγια να πω για την περίπτωση μη σύναψη Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία της Μεγάλης παρασκευή θα εξακολουθήσει να ισχύει και το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι συνεγγυητή αυτή τη συμφωνίας. Και θα πρέπει να σεβαστεί το πνεύμα και το γράμμα τη Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να διαθέσει και επιπλέον πόρους στην Ιρλανδία και τεχνικού και οικονομικού για να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε επιπλέον πρόκληση. Οπότε ο σεβασμό τη Συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή θα είναι ο μύτο τη Αριάδη για να αποφύγουμε ένα σκληρό σύνορο. Αλλά μια και πρόκειται για το σεβασμό τη ενία αγορά, τη δική μα εσωτερική αγορά, αλλά και για το σεβασμό τη ε, βρετανική εσωτερική αγορά, θα πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Κάποιο είδου έλεγχοι θα πρέπει να εφαρμοστούν. Περί αυτού πρόκειται. Εδώ και μια διετία λοιπόν διενεργούμε αυτές τις διαπραγματεύσεις που εξακολουθούν να είναι αρνητικές διαπραγματεύσεις. Δεν έχουμε καμία προστιθέμενη αξία του Brexit. Κανεί, ούτε καν ο κύριος Φαράζ, ο παρακαθήμενος, δεν κατάφερε να μας αποδείξει την προστιθέμενη αξία του Brexit. Κανεί δεν κατάφερε να το αποδείξει. Είναι αρνητική λοιπόν η διαπραγμάτευση. Όλοι βγαίνουν χαμένοι, lose-lose. Κανένας δεν επωφελείται από τον Brexit. Ως εκ τούτου θα πρέπει με ευφυΐα να βρούμε μία συμφωνία και μία λύση για να περιορίσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της διαπραγμάτευσης και να ολοκληρώσουμε ε, το εγχείρημα αυτό το συντομότερο δυνατό. Γιατί, όπως είπαν και κάποιοι προλαλήσαντες, έχουμε τόσο πολλά να κάνουμε και πέραν του Brexit. Ε, για το θετικό πρόγραμμα που ανέφεραν ο κύριος Τούσκο, ο κύριος Κατάινεν, θα πει αργότερα. Αυτό μετράει και σε αυτό αυτό το πολιτικό μας ε, πρόγραμμα και το θετικό πρόγραμμα να ξεπεράσουμε αυτό το διαζύγιο που θέλουμε να το οργανώσουμε όσο πιο τακτικά γίνεται, να επικεντρωθούμε στο πολιτικό μας πρόγραμμα του πιο σημαντικού, της οικοδόμησης με το Μένο Βασίλειο και της σφυριλάτησης ισχυρής και βιώσιμης μακροχρόνιας σχέσης με μια χώρα που θα παραμείνει φίλος, σύμμαχος και εταίρος η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θέλω να πω εγκατακλείδη, ήταν μια πολύ σοβαρή απόφαση για να αντιμετωπιστεί αυτή η μερικές φορές απροσδόκητη κατάσταση στη Βουλή των Κοινοτήτων και να εκλάβεται αυτή την απόφαση ως την βούληση, την επιθυμία των Ευρωπαίων να μπορέσει το, το Ηνωμένο Βασίλειο κυρίαρχο να λάβει τις αποφάσεις του και να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επιλέξει τι θα αποφασίσει. Αυτό που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τη διπλή απόφαση ε, τις δύο ημερομηνίες δηλαδή, τον Απρίλιο και τον Μάιο, προβλέπει ακριβώς τη δυνατότητα που ανοίγεται για το Ηνωμένο Βασίλειο να αναλάβει τις ευθύνες του, να υπομειστεί τις ευθύνες του. Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η χώρα που θέλει να αποχωρήσει, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνε του, να αποφασίσει για το μέλλον του και φυσικά να υπομειστεί τι συνέπειε των αποφάσεών του. Γιατί κυρίες και κύριοι, αυτή η διαπραγμάτευση δεν ήταν εμπορική διαπραγμάτευση. Δεν ε, είναι δοσοληψίες και παραχωρήσεις από όλα τα συμβαλωμένα μέρη. Είναι μια διαδικασία εξόδου. Το, Ευρω... το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να αποχωρήσει από την ενιαία αγορά, από την Τελωνιακή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβει τι ευθύνε του και να αντιμετωπίσει και τι συνέπειε. Παρόλο που, όπω είπε ο κ. Τουσκ, όλα είναι ακόμη δυνατά μέχρι τι 11 Απριλίου. Πάντω, οποιαδήποτε επιλογή θα έχει συνέπειε και θα πρέπει τι συνέπειε να τι επομιστεί το Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνοντα ευθύνη και αναλαμβάνοντα την κυριαρχία του. Γιατί αυτή τη η δυνατότητα διανοίγεται με την απόφαση και τη διπλή ημερομηνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Και εμεί σα ευχαριστούμε, κύριε Μπαρνιέ. Επόμενο ομιλητή, ο Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Κατάινεν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Παρότι η συζήτηση έχει εστιαστεί σχεδόν αποκλειστικά και μόνο στο θέμα του Brexit. Δεν θα περιοριστώ μόνο σε αυτό, γιατί ο κύριο Μπαρνιέ, ο βασικό μα ε, και κύριο διαπραγματευτής, θα εξήγησε πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα εγώ να σχολιάσω κάποια άλλα θέματα που επίση συζητηθήκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο ε, στην βιομηχανική πολιτική και στη σχέση με την Κίνα. Πολύ σύντομα, όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική, έχει ήδη συσταθεί μια ομάδα εργασία, ομάδα εμπειρογνωμόνων που ασχολείται με το μέλλον τη ε, βιομηχανική πολιτική. στην Ευρώπη με στόχο το 2030. Αυτή λοιπόν η ομάδα ήδη δουλεύει εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Εγώ συμπροεδρεύω μαζί με την Επίτροπο Μπιετσκόφσκα και θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν το έγγραφο ε, θα διατεθεί στο επόμενο κοινοβούλιο. Ο στόχος είναι να εντοπίσουμε τα κέρια σημεία για το πώς μπορούμε να εξυγχρονίσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε ήταν η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις προτάσεις μας και σε μεγάλο βαθμό τις στήριξε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα είναι στρατηγικοί εταίροι. Και οι στρατηγικοί εταίροι κατά κανόνα όχι μόνο μιλάνε μεταξύ τους αλλά κάνουν και συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτό το τελευταίο ε, πρόσφατα είναι λιγάκι προβληματικό. Συμφωνούμε σε πάρα πολλά με τις